Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ετιγκέρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ως κύριε εισηγητρία για το θέμα αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που είχα να συγκροτήσω μια έκθεση η οποία είχε πολλές φιλοδοξίες και πολλές συμβολές από τους συναδέλφους. Νομίζω ότι καταδεικνύει την τωρινή κατάσταση της εργασίας της Επιτροπής μας και έχει και προτάσει για το μέλλον. Ο στόχος της έκθεσης είναι η περαιτέρω βελτίωση του έργου μας για τις αναφορές. Κάποιοι από εμά μπορεί να έχουν επικρίσεις σε σχέση με ορισμένε ε, ε, απόψεις για την ε, έκθεση αυτή αλλά αυτό <clears throat> είναι καλό, είναι θετικό. Δείχνει ότι υπάρχει μια πολυφωνία, δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα τομείς στους οποίους εμείς θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και εμείς θα κάνουμε όλα αυτά τα οποία θα μας φέρουν κοντύτερα στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ελπίζω θα οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικό έργο της Επιτροπής Αναφορών προς όφελος των πολιτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τις λεπτομερείς εξηγήσεις του και νομίζω ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών πολλών ανθρώπων. Χρησιμοποιώ λοιπόν και αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές μου γιατί ήταν πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις τους Μπέκερ, Αλμπιόλ, Εύη, Μπετσέρα, Μαριάς, Ρέντα. Όλους αυτούς θέλω να ευχαριστήσω και επίσης θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συντονιστές, συμβούλους, το προσωπικό της γραμματείας, που εργάστηκαν για αυτή την εργασία και τον κύριο Καμπεθόν Μπάιδο, Κύρκος Περές και την ε, βοηθό μου την κυρία Μπέρσκα. Παρά τις αρχικές ε, δυσκολίες και διαφορές μπορέσαμε να υποβάλουμε μια αξιόπιστη έκθεση για το μελλοντικό έργο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Πέρα της συζήτηση η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12, σε 2,5 λεπτά δηλαδή. Με άλλα λόγια διακόπτουμε μέχρι τις 12. Ευχαριστώ.